Συνάδελφοι, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε τις εξηγήσεις ψήφου, οπότε παρακαλώ όσοι δεν συμμετάσχετε να βγείτε από την αίθουσα. Και τώρα θα περάσουμε σε επεξήγηση ψήφου, αγαπητοί συνάδελφοι. Έκθεση για την υγεία των ζώων και για ένα λεπτό μπορεί να πάρει το λόγο η κυρία Μορβέη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ, κυρία Μορβέη, στο συγγνώμη. Κοιτάξτε, ε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την τάξη εδώ. Έχετε το λόγο κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι πολύ ταραγμένη. Δεν τολμάω να πω τίποτα. Να είναι το στόμα μου. Γιατί ανησυχώ βαθύτατα για το αν ο πρόεδρος Μάρτιν Σούρτς έχει προλάβει να πάρει το αεροπλάνο του. Πάει λέει στην ε, Βόρεια Κορέα να τους κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Βιαστικός, βιαστικός έφυγε. Ελπίζω να την πρόλαβε την πτήση του. Υγεία των ζώων λοιπόν και προστασία αυτής. Όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με γεωργική πολιτική, οικονομική πολιτική και εκβιομηχάνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιομηχάνηση γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποβαίνουν εις βάρος της ε, Υγεία των ζώων, πιστεύω. Βλάπτουν τις μικρές επιχειρήσεις. Καλύτερα θα ήταν να μεριμνούσαμε να προστατέψουμε καλύτερα την υγεία των ζώων. Ευχαριστώ και σε ένα λεπτό μόνο, παρακαλώ να γίνεται σεβαστός ο χρόνο, κυρία Γκίλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ υποστήριξα την έκθεση για την υγεία των ζώων, καθώς σημαίνει βήματα προοδευτικά προόδου για την χάραξη πολιτικής, την οποία εγώ βέβαια υποστηρίζω. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους δικούς μου ψηφοφόρους που θέλουν να προστατεύεται η υγεία των ζώων, θέλουν μια σαφή στρατηγική. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπογραμμίσουμε το πλαίσιο δράσης της εκθέσεως κυρίως για τις λοιμώδεις επιζωτίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Εν προκειμένου καλωσορίζω την τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας λέει ότι αγωνίζεται για την προστασία της υγείας και προγωγή της υγείας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια όλο καλή έκθεση που γίνεται προς την ορθή κατεύθυνση και σας ευχαριστώ. Κύριε Χάραν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια από τις πιο φλιβερές τάσεις στην περίοδο που ζούμε είναι το να χρησιμοποιεί κανείς την ομοθεσία για λόγους ηθικούς, ηθικού κύρους, για να δείχνετε καλός άνθρωπος που είναι. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει κάτι να ε, επισημάνουμε, ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της προστασίας της υγείας των ζώων και της επικράτησης επιζωτιών, που άλλωστε καταδεικνύει και η έκθεση, με την μαζική ε, γεωργική παραγωγή των τελευταίων δεκαετιών έχουμε απλώς εξασφαλίσει ένα περιβάλλον ε, αντισηπτικό για να μην διαδίδονται οι λοιμώδεις επιζώτιες. Ωστόσο, με το που θελήσαμε να έχουμε ένα πιο φυσικό περιβάλλον για τα ζώα, άρχισαν να διαδίδονται και αυτές οι επιζωτίες και ακριβώς εδώ είναι η δυσκολία. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ευημερία και υγεία ταυτόχρονα. Οι τοπικές αρχές πρέπει να σε θέση να τα αποφασίζουν αυτά. Ερετές τοπικές αρχές. Ευχαριστώ και τώρα προσοχής ο κύριος Πόσπης. Και σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα τον ε, κανονισμό καθώς κάθε φορά υποστηρίζω νομοθεσία η οποία βαίνει προς όφελος της υγείας των ζώων. Πρόκειται λοιπόν για μια αρχή που θα πρέπει να υιοθετούμε πάντα και να έχουμε και μέτρα αντιμετώπισης των επιζωτιών. Δεν υπάρχουν ωστόσο διαδικασίες πάντοτε ικανοποιητικές. Με χαρά και ανακούφιση βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει στις δηλώσεις της την ε, ε, προστασία των ζώων και την ε, ευημερία τους. Ήταν καλό να κοιτάξουμε θέματα προστασίας της ευημερίας των ζώων με μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον και ασφαλώς υπάρχουν πτυχές άλλες που είναι λιγότερο απτές ίσως. Μίτσι. Πρόεδρε, ευχαριστώ τα τελευταία χρόνια. Η πρόοδο στην ευημερία των ζώων και η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχουν χάσει το ρυθμό του. Αλλά σήμερα σημειώνεται σημαντική πρόοδο με την υιοθέτηση σχετική νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Μπορεί η νομοθεσία αυτή να μην αφορά συγκεκριμένα την νομοθεσία των ζώων, αποτελεί όμω ορόσημο στην ευημερία αυτών και μπορεί να αποτελέσει και ένα ε, σημείο καμπής για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν τα κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα για την υγεία και την εφημερία των ζώων, ο κτηνοτρόφος, ο εκτρέφων ζώα θα έχει κανόνες ε, ορθής εκτροφής για να μην ε, υποφέρουν τα ζώα και να μην κινδυνεύει η υγεία τους. Επίσης θα πρέπει αυτές, αυτοί οι κανόνες να ισχύουν για όλα τα ζώα, είτε είναι οικόσιτα εκτρεφόμενα, είτε ε, αδέσποτα. Πρέπει να έχουμε σαφεί ευρωπαϊκέ δραστηριότητε για να εξασφαλίσετε για όλα τα ζώα ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία και σα ευχαριστώ. Thank you, Κύριο Μάμικιν, ένα λεπτό. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μιλούμε για την αντιμικροβιακή αντίσταση και μέτρα για την αντιμετώπιση της. και για μια πιο προσεκτική χρήση των αντιβιωτικών και άλλων σχετικών φαρμάκων. Πρέπει να γίνει μια καλή συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι μπορούμε να προωθήσουμε τη συλλογή των δεδομένων και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και για την υγεία των ζώων γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την υγεία των ζώων. Παρακαλώ, Πόλτσακ. Το θέμα δεν είναι να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τα ζώα. Στο ρωμαϊκό δίκαιο τα ζώα ήταν πράγματα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Πρέπει να τα θεωρούμε ζώντες οργανισμούς που υποφέρουν, που αισθάνονται και που είναι τμήματα του περιβάλλοντός μας. Ε, όμως εδώ δεν πρόκειται μόνο για τα δικαιώματα των ζώων, κατ' επέκταση ε, αφορά τα δικαιώματα των ε, συμπολιτών μας, γιατί τα καταναλωτικά δικαιώματα είναι τμήμα αυτού του μεγαλύτερου οικοσυστήματος, εντός του οποίου τα δικαιώματα των ζώων θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά. Αντίσταση στα βιωτικά τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται μαζικά στα ζώα είναι προβληματική υπόθεση και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε αύριο. Ευχαριστώ. Ε, θα ψηφίσουμε μάλλον αύριο, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Στάκουλα. Θέλω να ε, ευχαριστήσω τους εισηγητές. Έκαναν εξαιρετική δουλειά σε αυτή την έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Σημαντικό το θέμα της ευημερία των ζώων και εδώ πρώτη φορά συνδυάζεται η ευημερία των ζώων με την ανθρώπινη ευημερία. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο ανεφέρθη ε, είναι η μείωση της κρίσης αντιβιωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε τα αντιβιωτικά να είναι αποτελεσματικά στο μέλλον Τα υπολείμματα των αντιβιωτικών στο ζωικό κρέας έχουν αποδυναμώσει και την επίδρασή τους στους ανθρώπινους οργανισμούς. Και εφόσον ζούμε σε οικονομία της αγοράς, σε ενιαία αγορά, είναι σημαντικό να φροντίσουμε για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων κατά συνέπεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Εγώ υποστήριξα αυτή την έκθεση και θέλω να επενέσω την Επιτροπή Άγρη καθώς και όσοι συνεργάστηκαν στο τριμερί. Πρέπει όντως να υπάρξει προληπτικός έλεγχος των επιζωτιών που είναι μεταδοτικές για τα ζώα αλλά και για τους ανθρώπους, όχι μόνο προς χάρη της, υγείας των, της ευημερίας των ζώων αλλά και προς χάρη της ανθρώπινης υγείας. Θα πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε ασθένειες και πιθανές τάσεις και να διατηρήσουμε και να παρακολουθούμε τις νομοθεσίες σχετικά με την ευημερία των ζώων. Αποτέλεσμα αυτών βέβαια θα πρέπει να είναι η μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών στα ζώα και άρα βελτίωση της ποιότητας ζωής για τα ζώα. Όσον αφορά την Ιρλανδία, εμείς εξάγουμε 40% της παραγωγής μας, κυρίως του βόηου κρέατος και η εκθεσευτή μας βοηθά στο να διατηρήσουμε τις υψηλές μας προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και περνάμε στην έκθεση Ταραμπέλα. Το λόγο έχει η κυρία Μορβάη. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σημαντικό θέμα είναι η διανομή προλαχανικών σχολικά ε, συγκροτήματα κυρίως προερχομένων βέβαια από τις ε, τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται όμως αυτή η τοπική παραγωγή δεν τους υποστηρίζουμε επί περιπτώσει δεν την κάνουν υποστήριξης ε, ούτε ο Πορώνης δεν βλέπουμε καλά καλά να υπάρχουν. Δεν ε, λειτουργηγούν οι τοπικές κοινωνίες αφού έχει καταστρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την δραστηριότητα. Και το τοπίο βέβαια της Ουγγαρίας. Μια μικρό υποστήριξη μπορεί να είναι αυτή η διανομή προλαχανικών στα σχολεία. Η κυρία Γκίλ έχει το λόγο. Στήριξα την έκθεση αυτή και είχα πει και στα σχόλιά μου προ τον εισηγητή ότι θεωρώ ότι είναι καλή έκθεση. Θα πρέπει βεβαίω για αυτό το πρόγραμμα να εγκρίνει τον προπολογισμό και το Κοινοβούλιο για το διάστημα 2017-2018. Έχουμε μεταφέρει τα απαραίτητα κονδύλια για να αυξήσουμε το την ετήσια προκοδότηση του προγράμματος αυτού, αλλά ε, αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ε, ήδη από το 1999 είχε αποβάλει τροπολογία για την πρωτοβουλία για το γάλα στα σχολεία και καλωσορίζω όλος ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εδώ προβλέπονται διατροφικές εναλλακτικέ ε, από τα αμφιγεινά σνακ και αναψεκτικά που καταναλώνουν σήμερα τα παιδιά. Εδώ λοιπόν αυτό είναι σημαντικό και για τους γεωργούς και τα παιδιά μας και επίσης μια πολύ καλή ε, συμφωνία για τον Βρετανό φορολογούμενο. Είναι άλλο ένας λόγος να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στα 17 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, ε, όχι για πολύ ακόμα, ιδίω αν πετύχει το δημοψήφισμα, αλλά ε, τα χρόνια αυτά ε, λόμπι γίνεται για το γάλα στα σχολεία και από του ε, και από του τους ε, εκπαιδευτικού, αλλά και από του γεωργού. Εδώ μάλιστα λέγεται ότι έχουμε πολύ κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων στη δίαιτα, στο θητολόγιο της διατροφής. Αλλά μου λένε μην τους ε, λέτε τι να κάνουν στο σχολείο, αφήστε το ότι τα κανονίζουν μόνα του, μόνοι τους. Τι συντονισμός είναι αυτός, γιατί αυτό το είδος το θέμα καθορίζεται α, για, έξι, για μισό εκατομμύριο πολίτες. Ε, για μισό δισεκατομμύριο πολίτες. Ποιος ο λόγος Βεβαίως υπάρχει απόσταση μεταξύ των τοπικών αρχών, των κυβερνήσεων της κάθε χώρας και της, των αποφάσεων που παίρνονται στις Βρυξέλλες. Αλλά αυτό συμβαίνει για να προωθούνται τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Ευχαριστούμε ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ που υπερψήφισα την έκθεση αυτή για την ε, διανομή μπανανών οπροκυπευτικών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ε, γιατί ο στόχο είναι να εγκριθεί ένα καλύτερο διαιτολόγιο, ένα πιο ισορροπημένο διαιτολόγιο για του νέου. Εδώ. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα θα είναι μέρος του όλου συστήματος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι καλύτερης ποιότητας και φυσικά. Ο νέος κανονισμός που θα αρχίσει να ισχύει από τον Αύγουστο του 2017 δίνει έμφαση στους τοπικούς παραγωγούς και στην παραγωγή εγκύτητας. Τα χρηματοδοτικά μέσα αυξάνονται κατά 20 εκατομμύρια, το ίδιο και τα παιδιά που βρίσκονται σε λιγότερο ευνοούμενα κοινωνικά στρώματα. Αυτά θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο. Πώς Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, στήριξα την έκθεση αυτή και ε, τον κανονισμό, διότι νομίζω ότι είναι σοβαρό να ασχοληθούμε με, την, με το διπλολόγιο των νέων, διότι οι καταχρήσεις και το, η γενική διατροφή είναι πρόβλημα σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η καλύτερη διατροφή στα σχολεία θα καθορίσει μελλοντικά τις επιλογές των ειδικών αυτών. Δεν μπορούμε βεβαίως να αναγκάσουμε τα παιδιά, αλλά μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτά τα προϊόντα για το γεγονός του, θα, του κατά πόσο θα βοηθήσουν οι ενισχύσεις. Και αν και στο παρελθόν οι επιδοτήσεις βοήθησαν και επέτρεψαν στους νέους να επιτρέπονται καλύτερα ή του γεωργού. Νομίζω ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα πρέπει να κοιτάξουμε προ το παρελθόν και να καταλάβουμε ότι το σύστημα παροχή βοήθεια ήταν αποτελεσματικό και καθόρισε τι καλύτερες επιλογές διατροφή στα σχολεία, γιατί πραγματικά χρησιμοποιούνται από τα σχολεία. Ευχαριστούμε κύριο Μάμικιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η υγεία των παιδιών μας και η εκπαίδευση στα σχολεία είναι ραχοκοκαλιά τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Εάν δεν υπάρξουν παιδιά, δεν υπάρχει μέλλον. Εγώ συμφωνώ με τη χρήση περισσότερων απορροκεπευτικών και γάλακτος και μπανανών στα σχολεία. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε ενεργά να στηρίξουμε και τους γεωργούς μας. Είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως η δική μου, την Λετωνία που έχει υποφέρει πολύ μετά την πρόβλεψη του εμπάργου κατά της Ρωσίας, να ενισχυθεί τα νοπά απορροκυπευτικά είναι Πολύ καλύτερα για τη διατροφή των παιδιών από τη λόγου χάρη τα πατατάκια. Εδώ λοιπόν αυτές οι επιδοτήσεις μπορούν να φτάσουν τα 26 εκατομμύρια για όλα τα σχολεία και νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σύστημα. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Πόλτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε ε, για το λόγο. Αυτή η ιστορία δεν είναι μια ιστορία που μπορούμε να τη δούμε ε, ως άσπρη μαύρο. Εδώ κάποιες ε, τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Και εγώ διερωτήθηκα αν έπρεπε να υπερψηφίσω να καταψηφίσω αυτή την πρόταση. Εν τέλει την υπερψήφισα, διότι σε αντίθεση με το περσινό ψήφισμα, στην του μορφή του, υπήρξε μεγάλη μετατόπιση στην ε, Δημοκρατία της Τσεχίας έχουμε 3.000 σχολεία και 60.000 άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα για τα σχολεία και τη διατροφή τους. Ε, είναι πολύ πετυχημένο. Δεν λέω ότι όλα τα προϊόντα είναι αναγκαστικά τα πιο υγιεινά, όμως αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα διάφορα σνακ, την κοκακόλα που καταναλώνουν κατά κορών τα παιδιά, είναι, που είναι σίγουρα ανθυγιεινά, έστω το ζαχαρούχο γάλα, έστω κάποια άλλα προϊόντα, είναι σαφώς λιγότερο βλαβερά λιγότερα επιζήμια για την υγεία. Εδώ λοιπόν αυτή την συμπεριφορά καλό να την καλλιεργήσουμε μεταξύ των νέων αντί να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες εκ των υστέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή με βρήκε σύμφωνη διότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι σημαντικά για τη Σλοβακία. Βάσει των στατιστικών, τα σλοβακικά νοικοκυριά έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση γάλακτο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, Σλοβακία, το πρόγραμμα για, τα, για το γάλα στα σχολεία υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε το 2004 έχει επιτρέψει στα παιδιά και τους γονείς τους να αγοράζουν γαλακτοκομικά προϊόντα σε καλύτερες τιμές ενώ πολιτήρια, αυτόματε μηχανέ πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων, χάρη σε αυτό το σύστημα έχουν εγκατασταθεί σε πολλά σχολεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, απορροκυπευτικών και μπανανών καταθύνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η διαφοροποιημένη κατανάλωση προϊόντων και οι αλλαγέ στι διατροφικέ συνήθειε είναι μέρο τη όλη πολιτική μα μέρημνα για τη δημόσια υγεία. Και βεβαίω είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε κύριο Στάκουλας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον συγκεκριτή, τον κύριο Τραμπελά. Υπερψήφισα την έκθεση. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι η κατεξοχήν αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή, όμω είναι ένα σημαντικό θέμα. Και καλό είναι να ασχολούμαστε με ζητήματα δημόσια υγεία, όπω το τι καταναλώνεται στη διατροφή των σχολείων. σω οι διαφορετικέ χώρε διοργανώνονται με διαφορετικό τρόπο στο τι τρώνε. Όμω είναι σημαντικό να αναφερθεί. Είναι ζωτική σημασία για τη δημόσια υγεία, όπω προείπα. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε προβλήματα παχυσαρκία, διαβήτη Και οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών ε, πολλές φορές ε, τα κάνουν να πίνουν ε, ζαχαρούχα ροφήματα. Έτσι, η προσφορά απορροκυπευτικών και γαλακτοκομικών είναι πολύ σημαντική. Ο κ. Χάναν είναι πολύ επικριτικός κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φαίνεται να ε, μην θέλει να παραμείνει και να μην ακολουθεί τον Πρωθυπουργό του, τον κύριο Κάμερον, που έκανε μια μεταστροφή πλήρη. Τέλο πάντων, δεν θα πάνε αναγκαστικά τα πράγματα. Σα ευχαριστούμε, κύριε Χάναν, ούτω ή άλλω. Ο κύριο Κέλλη, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, υπερψήφισα την έκθεση γιατί πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι θετικό. Παρέχει διατροφικέ εναλλακτικέ στα ε, παιδιά στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη και είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτή, αυτά, τα προϊόντα, εφόσον παρέχονται, θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να αυξηθεί η κατανάλωση γαλακτοκομικών και προεκπαιδευτικών μεταξύ των παιδιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, καλλιεργούνται προϊόντα που είναι και επιλέξιμα για επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν τα προκυπευτικά, τα γαλακτοκομικά και οι μπανάνες, αλλά και άλλα προϊόντα όπως ξηρή καρπή, γιαούρτια, ε, μπορούν επιτυχημένα να καλλιεργηθούν μεταξύ των παιδιών για να ε, υλοποιηθούν και συστάσει κατανάλωση αντικαρκυνικών προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να επηρεάσουμε όσο μπορούμε προ το θετικό, προς την κατεύθυνση τη διατροφική συνήθεια των παιδιών. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Έκθεση Φλέκινστον. Κυρία Στάιλερ έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, εγώ υποστήριξα τις εκκλήσεις των Βρετανικών λιμένων Δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει νομοθεσία που θα ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα για την περιοχή της Σκωτίας και τους λιμένες της. Χρειάζεται μια διαδικασία που θα επιτρέπει σε κάθε διαπραγματευτική ομάδα να μπορεί να εκφράσει και πάνω απ' όλα να γνωρίσει το Συμβούλιο το σύνολο θεμητών ανησυχιών και μελημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή τη φορά λοιπόν πρέπει οι εξαιρέσει που απαιτούνται για τους λιμένες της Βρετανίας να συμπεριληφθούν στη συμφωνία για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ Γκίλ. Η εκλογική μου περιφέρεια των Δυτικών Midlands ε, είναι μακριά από τη θάλασσα. Δεν έχει λιμένες. Αλλά πρέπει να λειτουργούν σωστά οι λιμένες για να μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται προσπάθεια εξυγχρονισμού των λιμενικών υπηρεσιών και δυστυχώ πάλι δεν τα καταφέραμε. Η επιφυλάξη μου σε σχέση με τι τελευταίε αυτέ προτάσει είναι ότι δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν την ποικιλία εικόνα που παρουσιάζει ο λιμενικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και δεν έχουν μπορέσει να περιορίσουν, να συγκρατήσουν τι ε, περιβαλλοντικέ συνέπειε Επίσης το δικαίωμα στην ε, απεργία και πιθανές συνέπειες νομικού χαρακτήρα για τα συνδικάτα. Πρόκειται λοιπόν για ένα αμβλή εργαλείο. Κάποια στοιχεία της συμφωνίας μπορεί και να υποβαθμιστούν ακόμη περισσότερο στη διαδικασία του τριμερού διαλόγου και γι' αυτό όπως και λυπή συναδελφοί από τους εργατικούς καταψήφισα την έκθεση. Ευχαριστώ. Χάναν. Ακριβώς αυτό δείχνει γιατί θα ήταν καλύτερα να ήμασταν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπω δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, οι, ιδιαιτερισμοί της χώρας μας. Πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί ότι είναι διαφορετικά τα λιμάνια και δεν μπορούν να βρίσκονται σε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, δεν μπορούν να ε, επιδοτούνται οι Βρετανικοί λιμένες. Αντιθέτως παράγουν ε, κέρδος για το ε, Υπουργείο των Οικονομικών για τον Εθνικό Κορβανά μπορεί λοιπόν να υπάρχουν λιμάνια που μπορεί να βρίσκονται σε κάποιες ισότιμες σχέσεις όπως το Ρότερνταμ και η ε, Αμβέρση, παραδείγματι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι για όλα τα λιμάνια της Ευρώπης ισχύουν ήδη συνθήκε. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικών λιμένων. Γιατί δεν εξαιρούνται αυτοί, διότι απλούστατα όλη αυτή η υπόθεση έμεινε όμοιρο στα χέρια των κρατικών ενισχύσεων και της αντιπαράθεσης της Επιτροπής με το Κοινοβούλιο. Και εν τέλει, ένα σημαντικό, ένα σημαντικός κλάδος μένει ε, όμοιρος στα χέρια των μεγάλων συμφερόντων. Ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την πρόταση για τους λιμένες. Λίγα ήταν τα, τα ωφέλη για τους εργαζομένους ή το περιβάλλον δεν μπόρεσε δηλαδή να αξιοποιηθεί ευκαιρία για καλύτερες ε, διατάξεις σχετικέ με την απασχόληση και το περιβάλλον. Οι εργατικοί θα ε, συνεχίσουν να εργαζόμονται με τα συνδικάτα για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο αυτή η νομοθεσία. Με όλες τις ε, ιδιαιτερότητες του Ηνωμένου Βασιλείου και τη σχέση του με την ιστορική ε, αγορά πρέπει να θυμόμαστε ότι ακριβώς εάν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα σημάνει ότι δεν θα έχουμε φωνή, δεν θα ακουγόμαστε, δεν θα έχουμε ψήφο. Ως χώρα λοιπόν αλλά και ως περιφέρεια πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι απόλυτα ζωτική σημασία να μείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο για τις εργασίες, την απασχόληση, τα δικαιώματα, αλλά και για το μέλλον των λιμένων μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αν δεν σπάσει, μην το κολλάς, λέμε στα αγγλικά εμείς με τη σοφία μας. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν το ακούει για η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρώτες, πρώτοι λιμένες και σε παροχή υπηρεσιών και σε αποτελεσματικότητα σε όλο τον κόσμο. Και άρα πρέπει η αξιοσύνη να επενεθεί, όχι να υποβαθμιστεί για να εξασφαλιστεί ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Μα δυστυχώ αυτό ακριβώ πράττει ο σχετικό κανονισμό. Και πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα νομοθεσία κουβέρτα, η οποία κινδυνεύουμε να δούμε να καταστρέφει του ευρωπαϊκού λιμένε. Γραφειοκρατία δηλαδή που σημαίνουν ότι τα λιμάνια της δικής μου εκλογικής περιφέρειας που έχουν με κόπο μεγάλο κερδίσει την ανταγωνιστικότητά τους θα βρεθούν πάλι στην γραμμή της αφετηρίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε, να συνεργαζόμαστε και με τα συνδικάτα και με τους εργοδότες για ένα καλό επίπεδο λιμενικών υπηρεσιών και σας ευχαριστώ. Ιστορικά ο αθλητισμός έχει να παίξει ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό απαιτείται μια ορθότερη διαχείριση της δραστηριότητας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει υπό εξέταση πρόσφατα τα συστήματα στήριξης των κάτω χωρών και της Γαλλίας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Και δεν θα, πρέπει να κάνουμε τη σύγχυση ανάμεσα στο μέγα λιμένα του Ρότερνταμ και ένα μικρό ψαράδικο λιμανάκι της Λετωνίας. Δεν ε, χωράνε όλα λοιπόν στο ίδιο καλούπι. Δεν θα πρέπει επίσης ε, να ξεχνάμε και το τι λένε τα συνδικάτα τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ενοποίησης των ρυθμίσεων. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο. Απαιτείται να υπάρχει αυστηρή μορφή ελέγχου στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Απαιτείται να υπάρξουν εγγυήσει για τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό και των λιμενικών δραστηριοτήτων. Δεν θέλουμε μονοπόλια, δεν θέλουμε λαθρεμπόρια. Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς προς όλες τις κατευθύνσεις και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη δική μου χώρα, την Ρουμανία. Έχουμε λιμένες στην Κωνσταντζα, στο Ιάσιο, στο Γαλάτσι και όλα εντάσσονται σε ένα ενιαίο δίκτυο με διαφάνεια, χωρίς μονοπόλια, με λογιστικούς κανόνες αυστηρούς και ξεκάθαρους. Όπως επίσης και διαδικαστικούς κανόνες διαφανείς. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ και εγώ. Εγώ θα υπερψηφίσω με την πολιτική μου ομάδα Τη συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει πολλά καλά στοιχεία, θετικά στοιχεία, μας οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια <clears throat> σε σχέση με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν και εγγυήσει για τους ε, εργαζομένους. Θα πρέπει να δούμε και τι συνέβη βέβαια στο COP21 και τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τις εκπομπές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον τομέα των εκπομπών οι λιμένες ε, δεν θα πρέπει να ε, διαφύγουν της προσοχής μας. Εμείς ε, έχουμε ένα σημαντικό λιμένα στην περιοχή μας, το Σάνον, Σάνον Φόιν, έναν βαθύτατο λιμένα σε σχέση με, άλλους, με άλλες ευρωπαϊκές λιμενικές εγκαταστάσεις και θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε σωστά. Ευχαριστώ. Κύριε Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πλαίσιο, το ρυθμιστικό που προβλέπετε θα έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις των αγορών γύρω από το θέμα των λιμενικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ανεξάρτητος μηχανισμός έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν αναφορές και οι αναφορές να εξετάζονται από ανεξάρτητους οργανισμούς. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η ιδέα της συνεργασίας του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί η απαιτούμενη νομική ασφάλεια η πρόεδρος λέει ότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στις οικονομικά και οικολογικά αηφόρες μορφές μεταφορών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε στην επόμενη έκθεση κατά πολέμηση της απάτης, η κυρία Μορβάγη. Όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες. Θεωρώ πολύ σημαντικό να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτό τον τομέα. Γνωρίζουμε από την εμπειρία μας μέχρι τώρα ότι και εδώ υπάρχουν προβλήματα όταν ε, ε, βλέπουμε ε, ότι παραδείγματο χάρη στη Ρουμανία η καταπολέμηση της απάτης είναι αντικείμενο κατάχρησης και εκμετάλλευσης για πολιτικούς λόγους. Δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω την έκθεση αυτή λόγω ακριβώς των ελλημάτων που υπάρχουν. Παρότι η έκθεση αυτή συνεισφέρει στο να καταπολεμήσουμε καλύτερα την απάτη. Θα είμαι πολύ αυστηρή προς όλους. Ένα λεπτό μόνο. Η καταπολέμηση της απάτης ήταν βασικός στόχος της Ένωσης για πολλά χρόνια. Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει τις προκλήσεις, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε δηλαδή τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη και των πολιτών μας. Η έκθεση τονίζει πως υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου πολλά και το δικό μου, η Βρετανία, πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μεγάλο κομμάτι των απατών που αντιμετωπίζει η Ένωση είναι στο επίπεδο κρατών μελών. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ετοιμάσει μία έκθεση κατά της ε, διαφθοράς. Αυτό είναι πρόσδεκτο. Θα πρέπει επίσης να περιλάβει τη μεθοδολογία των ε, ποσοστών σφάλματος στην Ένωση και στα κράτη-μέλη. Παράλληλα, ωστόσο, πρέπει να υπάρχει νομοθεσία για το, επί, για το μικρότερο δυνατό ε, για ένα κάποιο ελάχιστο ποσοστό προστασίας των ε, ατόμων που αποκαλύπτουν τις απάτες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω την έκθεση αυτή για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή περιγράφει πολύ σωστά τα προβλήματα τα οποία συναντάμε στην πράξη υπάρχουν συχνά παραβάσεις ε, της νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής και αυτό θέλω να επεξηγήσω. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων όταν δημιουργούμε ένα νέο γραφείο, μια νέα υπηρεσία, μια νέα εισαγγελική υπηρεσία αυτή η νέα εισαγγελία δεν θα βελτιώσει την καταπολέμηση της απάτης. Η απάτη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω των συστημάτων δικαιοσύνης του κάθε κράτους μέλους. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να αποκαλύψει και να καταπολεμήσει την απάτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με το 2013, το 2014 αυξήθηκαν τα ποσοστά απάτης κατά 36% και οι παρατυπίες κατά 48%. 16.000 υποθέσεις ε, προέκυψαν. Εξετάζοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την πρόσφατη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και τις δαπάνες του 2014, βλέπουμε ε, αύξηση αυτών των δαπανών. Μιλάμε λοιπόν για τεράστια ποσά και κατασπατάληση πόρων. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ε, είχαμε ζημία 120 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής για υποχρεωτική δημοσίευση όλων των εγγράφων με βρίσκει σύμφωνα. Ευχαριστώ. Η επόμενη έκθεση, Έκθεση Μίλνερ. Κυρία Μόρβαη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω περαιτέρω γιατί καταψήφισα την έκθεση αυτή. Απλώς θα αναφέρω μια μικρή λεπτομέρεια, εμβληματική. Κάθε πολιτική της Ένωσης, εξωτερική και εσωτερική, θα πρέπει να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες οι, όλα τα άτομα με οποιαδήποτε ταυτότητα να έχουν να κερδίζουν. Αυτό είναι οι αξίες της Ένωσης. Ας μου εξηγήσει κάποιος, υπάρχουν άντρες, γυναίκες, άλλες σεξουαλικές ταυτότητες. Πώς μπορούμε όμως στη διαδικασία λήψη αποφάσεων να προσέχουμε ιδιαίτερα την ταυτότητα, τις ανάγκες ατόμων, την ταυτότητα το οποίο δεν γνωρίζουμε επακριβώς. Δεύτερον, μιλώ για άτομα που, που κερδίζουν 300 ευρώ το μήνα. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό. Η κυρία Τζίλς, να τονίσω ότι ήταν σημαντικό το ότι είχαμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε τόσες πολλές ε, ε, εκθέσεις ε, σήμερα για θέματα της γυναίκας. Και νομίζω ότι το mainstreaming για, για τη διάσταση του φύλου είναι σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας, γιατί ξέρετε τα κράτη-μέλη αργούν στην υλοποίηση πολλών από τις συστάσεις μας. Αν δείτε τη, διαφορά, τη μισολογική διαφορά μεταξύ φίλου στα στοιχεία στη Βρετανία δείχνουν ότι υπάρχει μισολογική ανισότητα 9,4%. Οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής, της επαγγελματικής τους ζωής τους, κερδίζουν, οι γυναίκες κερδίζουν πολύ λιγότερα από τους άνδρες. Πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό, ώστε οι γυναίκες να κερδίσουν αυτό το κενό. Υπάρχει επίσης ε, μία μικρός αριθμός παρουσία γυναικών στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική και στον τομέα της πληροφορικής από όπου προέρχομαι εγώ. Η κυρία Φορέντζα, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας παρουσίασε την έκθεση αυτή και μας επέτρεψε να την ψηφίσουμε σήμερα 8 Μαρτίου. Μακρά η παράδοση της 8ης Μαρτίου, μαχών των γυναικών για τα δικαιώματά τους. Γνωρίζουμε πόσο πίσω ανατρέχει ο αγώνας αυτός. Είναι σημαντικό να, να χαράξουμε ένα άλλο σημείο προς την πορεία αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την πλήρη... Ε, αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΔ που στην Ιταλία δεν υλοποιείται ακόμα. Η έκθεση αυτή πάντως παρέχει σαφείς και αποφασιστικές ενδείξεις προς την σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο υπερψήφισα αποφασιστικά την έκθεση. Mr. Ο Μαμίκης, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά ακρίμα το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται ότι όσα ψηφίσματα και αν υιοθετήσουμε, εμείς δεν εξυπηρετούμε τις αρχές μας, ιδιαίτερα στον τομέα της ισότητας των φύλων. Η ισότητα των φύλων είναι ένα καθοριστικό, θα έλεγα, χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής της χώρας. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει οι αρχές αυτές να γίνονται σεβαστές θα πρέπει να υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές και θα πρέπει να πάρουμε σωστά παραδείγματα από διάφορες χώρες και οργανώσεις. Επί τη βάση των αρχών της έκθεσης την υπεψήφισα συνεπώς. Ευχαριστώ η κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι απορρίπτω το αίτημα να υπάρξουν περισσότερες αρμοδιότητες σε αυτήν την Επιτροπή, ε, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, γιατί θα την καταστήσει ανώτερη από τις άλλες επιτροπές. Δεν το θέλουμε αυτό. Οι γυναίκες δεν το επιθυμούν αυτό. Εμείς δεν θέλουμε έναν μόνιμο εισηγητή για τα θέματα του mainstreaming και τα θέματα ε, της ισότητας. Συνεπώς η πρόταση η οποία γίνεται στην ουσία είναι μια αεροπειρατεία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας από την σκοτεινή γραφειοκρατία. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να πω ότι δεν στηρίζω εν πάση περιπτώσει την πρόταση αυτή. Ο κύριος Γιούρεκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η αφαίρεση από την έκθεση αυτή της αναφοράς στην ισότητα των φίλων ε, σημαίνει ότι αγνοούμε για μια ακόμη φορά τα δικαιώματα των γυναικών, των εκατομμυρίων οικογενειών και εκατομμυρίων γυναικών που θέλουν να είναι σε θέση να αναθρέψουν τα παιδιά τους και θέλουν να αφιερώσουν τη ζωή τους στην ανατροφή των παιδιών τους. Αυτές είναι βασικές θεμελιώδεις αξίες για την ζωή των οικογενειών, των παιδιών, των εθνών και της Ένωσης και δεν μπορεί η Ένωση να δείχνει τέτοια περιφρόνηση για τα δίκαια των οικογενειών είναι προφανές ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υπάρξει αναφορές και για το τι θέλει το λόμπι των ομοφιλοφίλων. Έκθεση Χάινεμπολ, η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση είναι πολύ σημαντική πιστεύω και θέλω να τονίσω τους λόγους για τους οποίους την υπερψήφισα Σήμερα είχαμε μια συζήτηση που δείχνει πόσο επικίνδυνες ε, είναι οι μορφές ρετσισμού και ξενοφοβίας στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα μεταναστευτικό φαινόμενο όπου δεν μπορούμε να διακρίνουμε ετούντες, πρόσφυγες, ε, μετανάστες αλλά για άτομα που αναζητούν μια αξιοπρεπή ζωή. Το μεταναστευτικό φαινόμενο που βιώνουμε είναι πολύ διαφορετικό από τα προγενέστερα, όπου υπήρχε μια σημαντική παρουσία ανδρών. Τώρα έχουμε ένα φαινόμενο οικογενειακής μετανάστευσης, άντρες, γυναίκες, παιδιά που περνούν τα σύνορα. Είναι λοιπόν σημαντικό και η έκθεση το κάνει με σωστό τρόπο να αναλύσουμε... Ευχαριστώ. Μόρβαι, ένα λεπτό. θα σας αναφέρω το σημείο 13 της εξαιρετικά επικίνδυνης έκθεσης Hannibal. Μορφές, έμφυλες μορφές βίας και διακρίσεως συνιστούν δίωξη και πρέπει να αποτελέσουν σωσ... βάσιμους λόγους αναζήτησης ε, διεθνούς προστασίας στην Ένωση. Αυτό είναι το τρικάκι. Όλες οι χώρες προέλευσης των, της παρούσης εισβολής προς την Ευρώπη έχουν σημαντικές διακρίσεις κατά των γυναικών. Η διάκριση αυτή αποτελεί βάση για χορήγηση ασύλου, όπως ε, λέει η κυρία Χάνιμπολ. Κάθε γυναίκα δηλαδή έχει το δικαίωμα να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει απαιτητό δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Όλες οι πόρτες λοιπόν ανοίγουν, ανοίγει η Ευρώπη, ο καθένας μπορεί να έρθει στην Ευρώπη. Προσέξτε, είναι πολύ επικίνδυνη η έκθεση αυτή. Κύριε λέει ένα λεπτό. Πρόεδρε, είμαι υπερήφανη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει τη φωνή του να ακουστεί για μια αδύναμη ομάδα όπως είναι οι γυναίκες πρόσφυγες και συγχαίρω την συνάδελφα Μαρία Χάνιμπολ που φέρνει αυτή την έκθεση και ε, κατήρτισε την έκθεση για το Κοινοβούλιο οι γυναίκες πρόσφυγες ε, ήδη υποφέρουν διότι πρέπει να φύγουν από τις χώρες ε, όπου υπάρχει πόλεμος ε, και δυστυχία. Επειδή είναι γυναίκες υπάρχει επιπλέον και σεξουαλική εκμετάλλευση, βία και διακριτική μεταχείριση. Χρειάζονται μέτρα για την προστασία αυτών των γυναικών που είναι μητέρες ή κόρες. Οι διαδικασίες ασύλου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευάλωτο των γυναικών και χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν οι διακινητές και να οργανώνονται οι εγκαταστάσει υποδοχή υποδοχής κατά τρόπο ώστε να έχουν χωριστό, τόπο, ε, χωριστό χώρο διαμονής ε, και προσωπική υγιεινής. Χρειάζονται μέτρα για την προστασία αυτών των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκονζάλη Σπινά. Ευχαριστώ, Θυμάστε τον Donald Τάσκ την περασμένη εβδομάδα όταν μιλούσε για τους παράνομους μετανάστες που έμπαιναν σαν ε, τροκτικά στην ε, Ένωση. Ε, είναι μια προσβολή για χιλιάδες άτομα που φθάνουν στον, στις χώρες μας διοκόμενοι από τον πόλεμο. Δεν είναι παράνομοι οι άνθρωποι από τον Ιανουάριο. Το 55% των ατόμων που μπήκαν στην Ένωση είναι γυναίκες. Υποφέρουν από βία, εκμετάλλευση αντιμετωπίζουν κινδύνους υγείας. Είναι αναγκαίο να ανοίξουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να διευκολύνουμε την ασφαλή και νόμιμη είσοδο των ατόμων αυτών. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί αποτελεί ένα ακόμα βήμα για να δώσουμε έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύοντα τις ειδικέ ανάγκες των γυναικών. Είναι θεμελιώδες ωστόσο να έχουμε και μέτρα διακόπτη η ο κύριος... Είναι σαφές ότι ήδη από την αρχή του 2015 ένα πολύ με ψηλό ποσοστό αυτών που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι γυναίκες και παιδιά. Και τώρα οι γυναίκες και τα παιδιά έχουν φτάσει το 55% το 2016. Συνεπώς λοιπόν οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολεμικής σύγκρουσης. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτής της ευάλωτης ομάδας και γι' αυτό θα υποστηρίξω την έκθεση αυτή Νομίζω ότι υπογραμμίζει τα στοιχεία τα οποία χρήζουν υπογράμμιση και καλούμεθα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστούμε τα υψηλά επίπεδα προστασίας τα οποία έχουμε ορίσει. Η κυρία Ζαμπόρσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις που έγιναν για τις γυναίκες οι οποίες ζητούν άσυλο και προστασία. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες αυτές, ιδιαίτερα οι μητέρες. Θαυμάζω τα αυτές τις γυναίκες και πρέπει να τους δώσουμε ε, μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα υπερψηφίσω όμως την έκθεση αυτή γιατί οι γυναίκες αυτές ε, είναι όμοιροι μια ιδεολογικής μάχης, μια ιδεολογικής πάλης. Υπάρχει επίσης και το θέμα το οποίο κοινικά τίθεται εδώ περί αμβλώσεων. Ε, νομίζω ότι αυτοί που ζητούν την ελευθερία των γυναικών θέλουν να πετύχουν ακριβώς το αντίθετο. Αλμπιόλ Γκουσμάν ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής γιατί σήμερα στις 8 Μαρτίου με χιλιάδες γυναίκες παγιδευμένες στα σύνορα πρέπει να θυμηθούμε την Ευρώπη των τυχών, την Ευρώπη του αποκλεισμού, την Ευρώπη που καταδικάζει τις γυναίκες που είναι συνένοχοι για την εκμετάλλευση και στον τομέα τον εργασιακό και στον σεξουαλικό τομέα τις καταδικάζει στις βόμβες. Οι γυναίκες δίνουν αγώνα λοιπόν και στην Ισπανία, στα εργασιακά και στην Παλαιστίνη και στο Σαχαραουή και στο Κουρδιστάν και στη Λατινική Αμερική εναντίον των εγκληματικών πρακτικών των πολιεθνικών όπως η συνδικαλίστρια ακτιβρίστια Κάσερες που δολοφονήθηκε στην Ονδούρα. Ευχαριστώ. Κλείνει η διαδικασία. Διακόπτουμε μέχρι τις 3.